μόνη της αυτό. Όμως εδώ έχουμε να κάνουμε με κάτι πολύ περισσότερο από την παροχή υλική βοήθειας. Η πυρκαγιά στην Παναγία των Παρισίων μας ε, κατέστησε απόλυτα σαφές ότι μας ενώνει κάτι πολύ πιο σοβαρό και πιο βαθύ από κείμενα συνθήκων. Έχουμε κάτι κοινό και το αναγνωρίζουμε αυτό όταν βλέπουμε τι μπορούμε να χάσουμε. Και όταν αντιλαμβανόμαστε ότι θέλουμε να το υπερασπιστούμε όλοι μαζί. Την προηγούμενη εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των 27 Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων σε συμφωνία και με την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου χορήγησε μια παράταση ευέλικτη της περίοδου που προβλέπει το άρθρο 50 έως την 31η Οκτωβρίου του 2019. Πρόκειται για μια παράταση η οποία επιτρέπει περισσότερο χρόνο, χορηγεί περισσότερο χρόνο και ευελιξία στην κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου για να βρει μια δέξοδο από την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή και ελπίζω να την αξιοποιήσει κατά το καλύτερο δυνατό τρόπο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένει ένα σαφές μήνυμα από το Ηνωμένο Βασίλειο για τα περαιτέρω. Και αν κυρωθεί η Συμφωνία Αποχώρησης, η περίοδος παράτασης αυτομάτως Λίγη την πρώτη ημέρα του μήνα που θα ακολουθεί την ανακοίνωση της κύρωσης και άρα από εκείνη τη μέρα θα έχει αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο. Πρέπει να είναι απολύτω σαφέ ότι δεν πρόκειται να ξανανοίξει η συζήτηση για τη συμφωνία αποχώρηση. Ωστόσο, προκειμένου να διευκολυθεί η διαδικασία αποχώρησης, οι 27 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διατεθειμένοι να ξανασυστήσουν την πολιτική διακήρυξη για τη μελλοντική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο, εφόσον προχωρήσουν οι θέσεις ε, του Ηνωμένου Βασίλειου. Την προηγούμενη εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο άλλαξε ε, λογική σε σχέση με τη χορήγηση μιας πιο ήπιας παράτασης ε, για το Ηνωμένο Βασίλειο στην χορήγηση μιας μακρύτερης παράτασης, χρονικά μακρύτερης δηλαδή, πράγμα το οποίο και εγώ προτιμούσα για να είναι πιο επικοδομητική. Αυτό επιτρέπει την διατήρηση κάθε επιλογής, δηλαδή και την κυρίωση της υφισταμένης συμφωνίας αποχώρησης και την, τον αναλογισμό των συνθήκων και της επιλογής του Brexit, εφόσον το επιθυμεί ο Βρετανικός λαός. Επίσης, ε, με την παράταση αυτή μπορεί να δοθεί έμφαση και σε άλλες προτεραιότητες εξίσου σημαντικές που έχουν να κάνουν και με τις εμπορικές συναλλαγές με το Ηνωμένο Βασίλειο, ε, με, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, Επίσης, ε, ξέρω ότι ορισμένοι μπορεί να έχουν διατυπώσει ανησυχίες πως το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να έχει παρελκυστική και παρεμποδιστική τακτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, από εδώ και εμπρό με την παράταση αυτή. Ωστόσο δεν θελήσαμε να ακούσουμε αυτές τις φωνές και τις κασάνδρες και ε, θεωρούμε ότι η στάση μέχρι τώρα του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν και θα συνεχίσει να είναι η στάση ενός υπεύθυνου ε, μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχουμε κανένα λόγο να θεωρούμε ότι κάτι μπορεί να αλλάξει. Επίσης αυτή η παράταση και αυτή είναι η τρίτη θέση μας, επιτρέπει να μην υπάρξει καθυστέρηση στην διαδικασία τη ολοκλήρωση του Brexit που θα κρατήσει περισσότερο από έξι μήνε. Δηλαδή θα έχουμε περισσότερη βεβαιότητα για τι επιχειρήσει και του πολίτε για την εξέλιξη του Brexit. Μία από τι συνέπειε αυτή τη συμφωνία είναι ότι τον επόμενο μήνα στον Ηνωμένο Βασίλειο θα δεξαχθούν ευρωεκλογέ. Πρέπει αυτή την προοπτική να τη μετωπίσουμε με σοβαρότητα. Τα μέλη, οι Βρετανοί βουλευτέ του ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με πλήρη δικαιώματα και υποχρεώσεις για, για αρκετούς μήνες τουλάχιστον μετά τις ευρωεκλογές και αυτό ήθελα να το αναφέρω σήμερα διότι ε, αντετάχθην στην ε, ιδέα που κυκλοφορούσε σε περίπτωση παράτασης στο Ηνωμένο Βασίλειο να τύχει μεταχείρισης δεύτερης κατηγορίας μέλους. Αυτό το απορρίπτω λοιπόν και σας παρακαλώ και εσάς, εάν τυχόν και ακουστούν τέτοιε ιδέες εδώ στο Κοινοβούλιο, να τις απορρίψετε ανεπιφύλακτα. Και γνωρίζω ότι και από τις δύο πλευρές της μάχης, από τις δύο όχθες της μάχης, όλοι μας, εγώ προσωπικώς, είμαστε εξαντλημένοι από αυτή την ιστορία και το καταλαβαίνουμε, είναι απολύτως κατανοητό. Πλην όμως αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία για να πει κανείς άντε ας το κλείνουμε το θέμα, γιατί κουραστήκαμε μόνο και μόνο. Όχι, πρέπει να συνεχίσουμε το Brexit να το αντιμετωπίζουμε με πνεύμα ανοιχτό και τρόπο πολιτισμένο, διότι ό,τι και να συμβεί το πεπρωμένο μας είναι κοινό, θα είμαστε πάντα συνδεδεμένοι και θέλουμε να παραμείνουμε στενοί φίλοι και εταίροι και στο μέλλον. Κατά την ε, σύνοδο κορυφής ένας από τους ηγέτες μας είπε ότι δεν πρέπει να ονειροπολούμε και δεν πρέπει να θεωρούμε ότι μπορεί να αναστραφεί το Brexit. Απάντηση δεν έδωσα εκείνη τη στιγμή. Σήμερα όμως και ενώπιον ημών θέλω να πω πως αυτή τη δύσκολη στιγμή στην ιστορία μας χρειαζόμαστε ονειροπόλους, χρειαζόμαστε όνειρα. Δεν μπορούμε να υποκύψουμε στην μυρολατρεία. Τουλάχιστον για μας που θέλουμε μια καλύτερη και πιο ενωμένη Ευρώπη. Αγαπητοί φίλοι, πρόκειται για τελευταία συνεδρίαση που θα συναντηθούμε σε αυτή σας την βουλευτική περίοδο. Ελπίζω να έχω τη χαρά να σας ξαναδώ, τους περισσότερους από εσά τουλάχιστον, μετά τις εκλογές. Σας ευχαριστώ. Thank you very much, Mr. President. Ευχαριστώ και τώρα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ζωάν Jean-Claude Juncker. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, χθε ήταν μια πολύ δυσάρεστη μέρα για όσου αγαπούν τη Γαλλία και το Παρίσι. Στη ζωή όλων μας, το Παρίσι δεν είναι ένα τυχαίο μέρος είναι μια πόλη όπου όλοι θέλουμε να πάμε για να ξαναρωτευτούμε. Και το να διαπιστώνουμε ότι το Παρίσι υφίσταται μια τραγωδία που δεν είναι μόνο αρχιτεκτονική, αλλά αφορά τη ζωή όλων των Γάλλων. Να βλέπουμε οι φωτιές να καταστρέφουν το εξωτερικό σύμβολο της δύναμης της Γαλλίας γιατί πάρα πολλοί επισκέπτονται την ε, Παναγία των Παρισιών, την Notre Dame. Όλα αυτά μας λείβουν ιδιαίτερα. Ε, ένα σημαντικό σύμβολο της Γαλλίας υπέστη μια σοβαρή πληγή και είμαστε όλοι μόνοι. Έχουμε όλοι πληγή από αυτό το γεγονός και εκφράζω την πλήρη συμπαράσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία ήδη διακήρυξε ότι θα βοηθήσει όλες τις προσπάθειες που κάνει ε, η Γαλλία, το Παρίσι, η Γαλλία, η Ευρώπη, όλοι επλήγημεν και εκδηλώνουμε την αλληλεγγύη μας με τους Γάλλους φίλους. Since uh, Από τότε που ολοκληρώθηκαν εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγώ ίδιος περιμένουμε να ολοκληρωθεί το Brexit. Βεβαίω πρέπει να εστιάσουμε και σε πολλά άλλα θέματα. Στο θετικό θεματολόγιο που έχουμε εντοπιό μα. Και γι' αυτό θέλω να είμαι πολύ σύντομο. Την προηγούμενη εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, έλαβε μία ε, ενιαία, ενωμένη και υπεύθυνη απόφαση για να παραταθεί η περίοδο εφαρμογή του άρθρου 50 μέχρι 31 Οκτωβρίου τρέχοντο. Αυτή ήταν μία αποδεκτή λύση για τρει λόγου. Πρώτα απ' όλα, και με τη στήριξη του σώματός σας εγκρίναμε όλα τα αναγκαία έκτακτα μέτρα και είμαστε έτοιμοι να υπάρξει, εάν υπάρξει συμφωνία, ε, ε, Brexit χωρίς συμφωνία, αλλά η Ένωσή μας δεν έχει να κερδίσει τίποτα από την ε, σοβαρή ανταραχή που θα προκληθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτοί που θα επωφεληθούν είναι αυτοί που είναι κατά της διεθνού συνεργασίας και θέλουν να υπονομεύσουν τη διεθνή τάξη. Και ποτέ ούτως ή άλλως δεν πρόκειται να διώξουμε ένα μέλος μας. Δεύτερον, προστατεύσαμε την ακυρεότητα και τη λειτουργία και του σώματό σα και όλων των θεσμικών οργάνων. Αν το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθεί να είναι μέλο τη 23 Μαου, τότε πρέπει να διεξαχθούν και εκεί ευρωεκλογέ. Αν δεν το κάνει και αν δεν έχει επικυρωθεί η συμφωνία αποχώρηση μέχρι τι 22 Μαου, η παράταση θα λήξει στις 31 Μαΐου. Αυτή είναι η κατάσταση από πλευράς ε, νομικής κατάστασης. Επίσης, διασφαλίσαμε ότι δεν χρειάζεται να συζητούμε το Brexit ε, κάθε 15 ημερών. Και δώσαμε στον Ηνωμένο Βασίλειο το χρόνο και το περιθώριο για να ξεπεράσει το αδιέξοδο. Όταν θα αρχίσει να ισχύει η συμφωνία αποχώρηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεργαστεί όσο γίνεται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπω κατά τη διάρκεια ε, των διαπραγματεύσεων για τον Brexit. Η πλήρη διαφάνεια των διαπραγματεύσεών μα και η στενή και αποτελεσματική συνεργασία με την ομάδα Brexit του Κοινοβουλίου ήταν η ισχύ μα κατά τι διαπραγματεύσει και θέλουμε αυτέ οι καλέ πρακτικέ να συνεχιστούν και κατά την εφαρμογή τη συμφωνία αποχώρηση. Οποτεδήποτε θα πρέπει να ληφθούν αποφάσει σε αυτή την λεγόμενη κοινή επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα φροντίσει να συμμετέχει πλήρω στο Κοινοβούλιο και θα λάβει ιδιαίτερα υπόψη τι απόψει του. Μάθαμε να προσέχουμε ιδιαίτερα αυτά που συμβαίνουν στην Βουλή των Κοινοτήτων του τελευταίους μήνε. Αλλά θέλω να είμαι απόλυτα σαφής για τον Brexit. Τίποτα δεν μπορεί να αποφασιστεί εναντίον των αποφάσεων αυτού του οίκου τη Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Τίποτα δεν μπορεί να αποφασιστεί για τον Brexit χωρί να ληφθούν πλήρω υπόψη οι θέσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κύριε Πρόεδρε, ε, και κύριοι, στι 31 Οκτωβρίου θα λήξει η νέα προθεσμία για μια συντεταγμένη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και αν δεν έχει επικυρωθεί από το Βρετανικό Κοινοβούλιο μέχρι τότε η συμφωνία αποχώρηση, θα υπάρξει ένα σκληρό Brexit που όλοι θέλουμε να αποφύγουμε. Φυσικά, το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να αποφασίσει επίση να αποσύρει την αίτηση αποχώρηση. Αυτό το είπε σαφώ στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αλλά αυτή δεν είναι η υπόθεση εργασία μου. Όπω επίση δεν είναι ότι θα υπάρξει καμία παράταση μετά την 31η Οκτωβρίου. Δεν είναι η υπόθεση εργασίας μου, ούτε αυτή. Δεν μου αρέσει αυτή η ημερομηνία 31 Οκτωβρίου. Κατά τα άλλα δεν μου αρέσει λοιπόν. Γιατί είναι η τελευταία μέρα της θητείας μου ως Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και δεν μπορεί να γίνει λοιπόν για αυτό το λόγο καμία νυχτερινή ε, συνεδρίαση, γιατί στις 12 η ώρα θα πρέπει να αποχωρήσω εγώ. Αλλά μπορεί να παραμείνει ο Ντόναλτ Τούσκ. Ε, έγινα πρόεδρος της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί ήθελα να επιταχύνω τις εργασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί θεωρούσα ότι έπρεπε να γίνουν περισσότερα για την κοινωνική Ευρώπη. Κάναμε περισσότερα, αλλά όχι επαρκή. Επίσης, ήθελαν να γίνουν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις της ε, Οικονομικής και Νομισματικής Ένωση. Θα ήθελα για τη χρηματοδότηση της επόμενης περίοδου 21-28 να είχαμε συμφωνήσει. Και δεν μπορώ να δεχτώ ότι πολλοί νέοι, οι πολλοί ερευνητέ, οι φοιτητέ που απολαμβάνουν ε, ε, ενισχύσεις από το έρασμος να ε, υποστούν τις συνέπειες του Brexit. Δεν τους αξίζει κάτι τέτοιο. Πρέπει να φροντίσουμε ούτω ώστε να μην απομακρυνθούν από την Ευρώπη. Τώρα προς τα που θα πάει το Ηνωμένο Βασίλειο αυτό θα το αποφασίσει το Λονδίνο. Και όσο νωρίτερα τόσο καλύτερα. Χαιρετίζω ιδιαίτερα το ότι η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση τώρα βρίσκονται σε ε, διαπραγματεύσεις. Αυτό το χαιρετίζουμε ως πρόοδο. Και ε, στο βρετανικό πλαίσιο βέβαια είναι πρόοδος, αλλά δεν είναι φυσιολογικό. Το ότι οι κύριες δυνάμεις τόσο αργά αποφασίζουν να συνοηθούν, αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Και χαιρετίζω το ότι επιτέλους τώρα γίνονται αυτές οι διαπραγματεύσεις. Το πότε θα αποχωρήσουν από το Ηνωμένο Βασίλειο Βρετανία είναι δικό του θέμα. Το πότε και το πώς. Και βεβαίως ε, συμφωνήσαμε για μια συμφωνία αποχώρησης ε, τον Νοέμβριο του 2018. Αυτό το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων του περασμένου Νοεμβρίου εξακολουθεί να ισχύει. Σε καμία ε, περίπτωση δεν θα επιτρέψουμε επιπλέον διαπραγματεύσεις πάνω στη συμφωνία αποχώρησης. Για την πολιτική διακήρυξη για το μέλλον ε, των σχέσεων, αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε, αν εκφραστεί επιθυμία. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, το Brexit δεν είναι το μέλλον της Ένωσης. Το μέλλον της Ένωσής μας είναι πολύ περισσότερο από το Brexit. Το Brexit δεν πρέπει να δυσχεράνει τις εργασίες μας για τις μεγάλες προτεραιότητές μας. Γι' αυτό το λόγο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε επί δύο αρχών. Πρώτον, όσο είναι μέλος του Ηνωμένου Βασίλειου, υπολογίζουμε ότι θα είναι υπεύθυνη, έντιμη η συνεργασία μαζί του. Είναι αρχή. Είναι βασική αρχή της συνθήκης που πρέπει να γίνει σεβαστή. Δεν ε, υπολογίζουμε, απαιτούμε να υπάρξει υπεύθυνη και έντιμη συνεργασία. Δεύτερον, δεν υπάρχει κράτο μέλο δεύτερη κατηγορία. Αλλά ένα κράτο μέλο θέλει να αποχωρήσει από την Ένωση, 27 άλλοι πρέπει να έχουν το δικαίωμα να συνεδριάζουν χωριστά για τα θέματα του μέλλοντο τη Ένωση. Δεν είναι αυτό καινοτομία. Το Δεκέμβρη του 1997 ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ω πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ξεκίνησε το Eurogroup κατά τη άποψη των Βρετανών, των Σουηδών, των Δανών και κάποιων άλλων. Το Eurogroup είναι μια περιορισμένη μορφή συνεδρίασης για όσους ενδιαφέρονται για την οικονομική οικοδόμηση της Ένωσης και την νομισματική. Είχαν το δικαίωμα να συνεδριάζουν και συνεδριάζουν και τα αποτελέσματα είναι ουσιώδη. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει στρατηγικές προκλήσεις στις οποίες πρέπει να ανταποκριθεί. Πρώτα απ' όλα, στο Σύμπιου το Μάιο θα συζητήσουμε τις στρατηγικές μας κατευθύνσεις για τα επόμενα χρόνια. Και κατόπιν έχουμε και το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, επί του οποίου επί της αρχής πρέπει να αποφασιστεί τον Οκτώβριο και πρέπει να εκλεγεί η επόμενη ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, του οποίου το εκλογικό σώμα είναι το μεγαλύτερο μετά από αυτό τη Ινδία. Και πρέπει να εκλέξουμε και μια νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να ορίσει τον επόμενο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Το μέλλον τη ενωσή μα έχει να κάνει και με τη θέση μα στον κόσμο. Γιατί έχουμε εμπορικέ συμφωνίε. Πρέπει να δούμε τις σχέσεις μα με του μεγάλου διεθνεί εταίρου μα, ιδιαίτερα με την Κίνα, με την οποία την περασμένη εβδομάδα είχαμε μια πολύ επικοδομητική συνάντηση κορυφή και τον ε, προσεχή Ιούνιο στην Όζακα θα στο G20, όπου θα συζητήσουμε μεταξύ άλλων για το μέλλον του παγκοσμίου εμπορίου. Όλα αυτά είναι πραγματικά πιο ουσιώδη από τα επεισόδια που σχετίζονται με τον Brexit. Η Ευρώπη συνεχίζει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να θυμίσω στους συναδέλφους ότι στη διάρκεια αυτού του Συμβουλίου εγώ επέμεινα για την αξιοπρέπεια του Κοινοβουλίου, για το ρόλο που έχει. Δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως ταξί και οι διαπραγματεύσει για το Brexit θα πρέπει να λάβουν υπόψη το ρόλο του δικού μας θεσμού. Νομίζω πως αυτό είναι για μας προτεραιότητα και πιστεύω πως μιλώ εξ ονόματος όλων των συναδέλφων γιατί είμαστε το πρώτος θεσμός ε, στη συνθήκη και ε, θεωρούμε ότι πρέπει όλα τα 28 κατημέλη να σέβονται το Ευρωκοινοβούλιο. Ευχαριστώ εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ο κύριος Γκονζάλε Πόνς έχει τώρα το λόγο. Θα πρέπει να πω τον πόνο που ένιωσα εχθές όταν έβλεπα να καίγεται η καθεδρική της Νότρε Ντάμ. Η πυρκαγιά αυτή μας έχει επηρεάσει όλους, αν ήμασταν Γάλλοι. Όλοι αισθανόμαστε θλίψη το ίδιο αποσβολωμένοι ε, και αδύναμοι και σήμερα το πρωί όλοι θέλουμε να ξεκινήσουμε την ανοικοδόμηση. Οι λαοί δεν αναπτύσσονται όμως κλαίγοντας μαζί, αλλά προχωρώντας μαζί. Και η χθεσινή πυρκαγιά της Νότριντά μας κάνει περισσότερο Ευρωπαίους, όχι επειδή κλάψαμε μαζί, αλλά επειδή μαζί θα ανοικοδομήσουμε την, ε, τον καθεδρικό ναό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προσφέρει οικονομική βοήθεια και τεχνίτες, όλους ε, όσοι είναι απαραίτητοι για να ξαναχτίσει χτιστεί ο καθεδρικό Ναό όπω χτίζονταν και στο παρελθόν ακριβώ οι καθεδρικοί ναοί, καλώντα όλου να συνεργαστούν για ένα τέτοιο ε, όραμα. Η χθεσινή πυρκαγιά έδειξε πω οι Ευρωπαίοι δεν είμαστε ποτέ μόνοι μα. Η Ευρώπη είναι η απάντηση στη φωτιά, στην καταστροφή, στον εγωισμό και στην φτώχεια. Γι' αυτό ε, χτες το βράδυ βλέποντας να καίγεται ο καθεδρικός ναός αναρωτήθηκα ακόμα μια φορά ε, μα γιατί θέλουν να φύγουν από εδώ οι Βρετανοί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια κοινότητα αξιών και αρχών. Εάν το, μας φαίνεται πως δεν λειτουργεί ε, θα πρέπει να τη μεταρρυθμίσουμε για να λειτουργήσει καλύτερα. Αλλά δεν φεύγεις, δεν φεύγεις γιατί οι αξίες είναι κοινέ, παραμένουν κοινέ και σε καμιά περίπτωση δεν είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Ό,τι και αν γίνει Τρία διδάγματα πρέπει να αποκομίσω από το Brexit. Πρώτον, ότι στην πολιτική δεν μπορεί κανεί να υποσύσχεται αυτό που δεν μπορεί να πραγματοποιήσει. Δεύτερον, στην πολιτική τα ψεύδη πάντοτε φέρνουν ε, απογοητεύσει. Και έπειτα, ε, ε, οι δεσμοί που χτίζει η ιστορία δεν μπορούν να καταλύονται μόνο και μόνο από, λόγω εγωισμού. Το Brexit είναι κάτι το αόριστο και χωρίς ημερομηνία. Για μένα η Ευρώπη είναι ολοκληρωμένη. Ε, δεν είναι ολοκληρωμένοι χωρί το Ηνωμένο Βασίλειο. Αν οι πολιτικοί οι Βρετανοί όμω δεν μπορούν να βρουν λύση, α δώσουν το λόγο πάλι στο λαό. Έπειτα η πυρκαγιά τη Νοτραντάμ μα δείχνει και πάλι ότι μιλάμε υπερβολικά πολύ για τον Brexit και πολύ λίγο για όλα τα υπόλοιπα. Λυπάμαι για την ε, ματαιοδοξία των Βρετανών πολιτικών. Όμως σήμερα η θλίψη για την πυρκαγιά της Νότροντάμα με καθιστά ακόμα περισσότερο Ευρωπαίο παρά η απογοήτευσή μου λόγω της ανικανότητας. Ευχαριστώ εκ μέρου τη της Συμμαχία των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ο κύριο Ούντο Μπούλμαν έχει το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα το πρωί ενωμένοι κοιτάμε και στρέφουμε το βλέμμα προς το Παρίσι. Και θέλουμε να πούμε είμαστε η Νότρο Ντάμ. Θέλουμε να πούμε Παρίσι δεν είσαι μόνο σου. Γαλλικέλα, ε, δεν είσαι μόνος σου. Έτσι εκδηλώνουμε εμείς την ε, Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη. Και με αυτό το πνεύμα της Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης οφείλω να συγχαρώ εσάς, Πρόεδρε Τάσκ, τους που αναλάβατε εσείς την ευθύνη να χορηγήσετε την παράταση στο Ηνωμένο Βασίλειο για το Brexit, γιατί έτσι αποφύγατε την κατάρρευση, την σύγκρουση. Ποιος θα την πλήρωνε την κατάρρευση αυτή, τον κατακριμνισμό αυτών, ούτε η πολιτική, ούτε κανείς άλλος από τους μεγάλους και ισχυρούς, αλλά οι πολίτες αυτοί οι οποίοι μπορεί, μπορούν να ελπίζουν μόνο στο να βρούνε μία καλή δουλειά στο ένα ή το άλλο κράτος, αυτό που τους επιτρέπει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα ανοιχτά σύνορα. Και παίξατε με τη μοίρα των πολιτών της χώρας σας. Το απέφυγαν λοιπόν χάρη στον πρόεδρο Γιουνκέρ, χάρη στον πρόεδρο Τούσκ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τους υπεύθυνου πολιτικούς που έλαβαν την απόφαση της παράτασης. Και θα ήθελα να σας ε, επικροτήσω επίσης πρόεδρε Τούσκ όταν ε, είπατε ότι έχει δικαιώματα όπως κάθε κράτος μέλος όσο παραμένει μέλος και αυτό ισχύει και για του βουλευτέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν μιλούμε για μικροκομματικά ζητήματα ή επιλογές. Μιλούμε για αξιοπρέπεια του κάθε ψηφοφόρου της εκλογικής περιφέρειας, του κάθε εκπροσωπουμένου εδώ και βεβαίως θα καλωσορίσουμε τους εκλεγμένους εκπροσώπους στο Ευρωπαϊκό, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το Ηνωμένο Βασίλειο και θα έχουν κάθε ε, δικαίωμα και υποχρέωση και στη δική μου την πολιτική ομάδα εντασσόμενη σε κάθε περίπτωση. Και είμαι πεπισμένος ότι και μετά την 31η Οκτωβρίου θα ανοίξει μια νέα συζήτηση στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα αποτελέσει το έναυσμα του τέλους του Brexit. Είμαι πεπισμένος γι' αυτό. Γιατί εν τέλει θα έχουν την ευκαιρία οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου να μιλήσουν, να εκφράσουν τη γνώμη τους. Το Κοινοβούλιο, το Βρετανικό, δεν μπορεί να λάβει απόφαση. Σε τέτοιε περιπτώσει είμαι πεπισμένο ότι πάντα, πάντα πρέπει κανεί να στρέφεται στην ετοιμιγορία του λαού. Και ό,τι είναι στραβό να βγει από τη συζήτηση. Να παραμείνει ό,τι είναι σωστό. Το take back control σημαίνει δίνουμε το λόγο στο λαό, όχι στο δρυμερή διάλογο. Και είμαι πεπισμένο για το ότι το Brexit δεν αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο. Το Brexit δεν αφορά καν μόνο όλους αυτούς που θέλουν να μείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Brexit σημαίνει πολύ περισσότερα πράγματα. Έχει να κάνει με τους Πούτιν, με τους Τραμπ, με τους Στίβ Μπάνον, με τους Σαλβίνι που προσπαθούν να καταστρέψουν αυτά που έχτισαν ο Ρομπέρ Σουμάν και ο Ζαμονέ. Αυτά τα οποία ο Νάουερ και ο Βίλι Μπραντ οραματίστηκαν όλα αυτά τα οποία είναι κοινά και αυτά για τα οποία ακριβώς και θα υπερασπιστούμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί αποτελεί τη σωστή απάντηση στα μεγάλα ερωτηματικά για το μέλλον. Και βλέπουμε ποια είναι η απάντηση και στη Φινλανδία την είδαμε και στη Σουηδία τη βλέπουμε. Οι άνθρωποι θέλουν να αντιμετωπίσουν τους ακραίους δεξιούς και ενώνουν τις δυνάμεις τους και ελπίζω να δώσει την αντίστοιχη απάντηση με αυτή που δίνουμε εμείς και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα εκεί όπου στην Ανδαλουσία ή όπου αλλού έχει περιφερειακή περιφερειακές, τοπικές, ευρωπαϊκές, εθνικές εκλογές και στην Ιταλία και αλλού ανάλογα με το με ποιον θα συμμαχίσει θα κρυθεί η απάντηση που θα δώσει Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι ότι τασόμαστε στην Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο μέλλον. Ευχαριστώ. Συντηρητικοί και μεταρρυθμιστές της Ευρώπης, ο κύριος Καμάλ. Κύριε Πρόεδρε, όταν βλέπει κανείς τις εικόνες ε, χθε που και εγώ ήταν η Νότρα Ντάμ, είναι, ε, σκέφτεται ότι πρέπει να αφήσουμε την πολιτική κατά μέρο. Όπου και αν είναι, από όπου και αν είναι κανεί Βρετανό, από την Ευρώπη, από τον υπόλοιπο κόσμο, όλοι εθλίβησαν βαθιά. Πριν από 25 χρόνια η γυναίκα μου σπούδαζε στη Γαλλία και για ένα διάστημα εργαζόταν στη, στο Παρίσι και επισκεφτήκαμε την Notre Dame που είναι ένα σύμβολο και την προηγούμενη εβδομάδα ξαναπήγαμε. Πήραμε φωτογραφίες. Σκεφτείτε τα εκατομμύρια που επισκέφθηκαν ε, αυτή την εκκλησία ανεξάρτητα από την πίστη τους είναι σύμβολο όχι μόνο του Πασιού αλλά της ιστορίας της Ευρώπης αλλά ολόκληρου του κόσμου. Και ναι μεν εγώ ε, δεν είμαι αυτή τη πίστεως αλλά συμμερίζομαι τον πόνο σας εδώ σε αυτήν την αίθουσα και ελπίζω όλοι να συνεργαστούμε είτε Βρετανοί είτε Ευρωπαίοι είτε από πέρα από την Ευρώπη για να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πανικοδομηθεί. Δηλαδή, πολλοί ελπίζαμε ότι δεν θα γινόταν αυτή η συζήτηση σήμερα και ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα έχει αποχωρήσει Στι 29 Μαρτίου ή ακόμη και την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά πρέπει να αντιμετωπίσουμε με την κατάσταση όπω έχει. Η Βρετανική κυβέρνηση είναι ακόμη δεσμευμένη να υπάρξει συντεταγμένο Brexit και αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ω να τον πιο σύντομα. Αυτό ο στόχο τη, ούτω ώστε οι λαοί και των δύο πλευρών να εστιάσουν στο μέλλον. Αυτό που ανέφερε ο Ζαν Κλοντ Γιούγκερ, το θετικό θεματολόγιο. Ωστόσο, καταλαβαίνω ότι η υπομονή σα ε, έχει φτάσει στα όρια τη. Και Πραγματικά αναρωτιέστε τι συμβαίνει στο Westminster. Αλλά η συμμετοχή στην Ένωση έχει προκαλέσει ε, διχόνοια στη χώρα μου σε πολλά, για πολλά χρόνια. Όχι μόνο στο δικό μου κόμμα, αλλά και στο κύριο κόμμα τη αντιπολίτευση. Και αυτέ οι διχόνοιε βλέπετε πώ εξελίσσονται και τι ρόλο παίζουν. Και πολλοί ρωτάνε γιατί δεν συζητήσατε τι διακομματικέ συναντήσει νωρίτερα. Και μπορεί να φαίνεται φυσιολογικό για ορισμένου από τι χώρε τη δική σα, αλλά δεν λειτουργεί έτσι το κοινοβουλευτικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου. Κοιτάξτε τη Βουλή των Κοινοτήτων, όπου τα δύο κόμματα ε, κάθονται το ένα απέναντι από το άλλο. Όχι στο πλάι, όπω εδώ σε αυτό το κοινοβούλιο. Από τη μία πλευρά είναι η κυβέρνηση, από την άλλη η αντιπολίτευση. Και αντί να προσπαθούν να φτιάξουν ε, συνεργασίε, είναι πολύ πιο αντιπαραθετικό το σύστημα. Οι συζητήσει αυτέ που γίνονται τώρα δημιουργούν, ε, δημιουργούν συναισθήματα άβολη κατάσταση και από τι δύο πλευρέ. και σε μένα τον ίδιο. Η απάντηση λοιπόν που δόθηκε την προηγούμενη εβδομάδα τη παράτασης δεν είναι ίσως η ε, απάντηση που ήθελαν όλοι, αλλά είναι μια προσπάθεια να επιδιωχθούν άλλε λύσει. και ελπίζω οι συνάδελφοί μου στο Westminster να μην χρειαστεί να πάρουν πολύ χρόνο. Η οικονομία μα, η πολιτική μα ζωή και η χώρα μα χρειάζονται βεβαιότητα. Στόχο στόχος μας πρέπει να είναι να βρούμε μια λύση που θα μα επιτρέψει να αποφύγουμε τη συμμετοχή σε ευρωεκλογέ. Ήρθε τώρα η ώρα για πραγματι... πραγματισμό, για ρεαλισμό. Α τα καταφέρουμε. Και κύριε Τούσκ, σα ευχαριστώ για την πιο επικοδομητική σα στάση την προηγούμενη εβδομάδα σε σχέση με κάποιε άλλε δηλώσει που είχατε κάνει στο πρόσφατο παρελθόν. Νομίζω ότι τα λόγια σα πριν από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου είχαν το σωστό τόνο. Ότι το θέμα δεν είναι να ε, ταπεινωθεί κανεί ή να υπάρξουν αλληλοκατηγορίε. Πρέπει να παραμείνουμε φίλοι για να προχωρήσουμε στο μέλλον με μια ε, μελλοντική εταιρική σχέση που να διαρκεί. Το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν ε, και σε προηγούμενες καταστάσεις σε δύσκολη θέση, αλλά ε, τα καταφέρνουμε πάντα και ελπίζω ότι και αυτή τη φορά θα τα καταφέρουμε. Και διαρωτώ με αγαπητοί συνάδελφοι, για να πω κάτι προσωπικό. Ίσως είναι η τελευταία μου ομιλία από αυτή την έδρα, σε αυτό το εμικύκλιο μετά από σχεδόν 14 χρόνια. Θέλω να πω ότι ε, είτε συμφωνούσαμε, είτε διαφωνούσαμε, είτε πανεκλεγείτε, ή θα αντιμετωπίσετε νέε προκλήσει. Σα ευχαριστώ όλου ε, για την ε, εργασία σα που συμμετείχατε σε αυτή την καταπληκτική εμπειρία και εύχομαι σε όλου σα καλή τύχη, ό,τι καλύτερο για το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Καμά. Ο επόμενος, ο πρόεδρος της ε, ομάδας των φιλελευθέρων, κύριος Γκίφερ Χόστατ. Κύριε Πρόεδρε, όπως και οι συνάδελφοι, και ο πρόεδρος Τούσκ και ο πρόεδρος Γιούνκερ να εκφράσω και εγώ τον πόνο μου για την τρομερή πυρκαγιά χθες βράδυ στο Παρίσι. Είμαι πεπισμένος ότι από κοινού θα ξαναχτίσουμε την Νότο Ντάμ των Παρισίων και θα είναι ακόμη πιο όμορφη με περισσότερη ακτινοβολία από ό,τι στο παρελθόν. Η Παναγία των Παρισίων της Γαλλίας είναι η Παναγία της Ευρώπης. Είμαι πεπισμένος. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Τούσκ. Ξέρω ότι το κοινοβούλιο μας δεν ε, συμμετείχε στην απόφαση που πήρατε την προηγούμενη Τετάρτη. Παρ' όλα αυτά, θέλω να σας προειδοποιήσω για το εξής. Για τις επιπτώσεις ε, της απόφασης που λάβατε την, την προηγούμενη εβδομάδα. Γιατί μέχρι τώρα υπήρξε ενότητα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενότητα των 27. Αλλά ενότητα και μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων. Συμβουλίου, Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή η ενότητα βασιζόταν στην εργασία του διαπραγματευτή μας. Θέλω να το υπενθυμίσω αυτό. Ο Μισελ Μπαρνιέ, τον οποίον θέλω να συγχαρώ για τη θαυμάσια εργασία του. Και αυτή η ενότητα, κατά τη γνώμη μου, κύριε Τάσκ, πρέπει να σας πω ειλικρινά, ότι διακυβεύεται τώρα. Αντί να στείλουμε την κυρία με πίσω στο Λονδίνο χωρίς καμία παράταση ή το πολύ με μια πολύ σύντομη, λίγες μέρες, μια εβδομάδα, της δώσατε ένα εξάμεινο. Ένα εξάμεινο. Ξέρετε πολύ καλά ότι στις 31 Οκτωβρίου δεν υπάρχει επαρκή χρόνο για να υπάρξει ουσιώδη αναθεώρηση του Brexit και επίση αρκετά μακριά η 31 Οκτωβρίου για να υπάρχει επίγουσα ανάγκη για δράση. Αυτές είναι οι επιπτώσεις. Βέβαια δεν ε, αποκαλώ την απόφαση αυτή βλακίες, όπως λέει ο κύριος Κόμπερν, ο οποίος ό,τι κάνουμε εδώ πέρα τα λέει βλακίες, αλλά εν πάση περιπτώσει φοβάμαι ότι θα συνεχιστεί η αβεβαιότητα και θα παραταθεί η αναποφασιστικότητα και φοβάμαι ότι θα εισαγάγει τα χάλια του Brexit σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα δηλητηριάσει τις επικείμενες ευρωεκλογέ. Περαιτέρω, φοβάμαι ότι... Ξέρετε, υπάρχει μια έκφραση στα Ολλανδικά. Θα κάνει το κοινοβούλιο μας, φοβάμαι, θα το κάνει σαν περιστερεώνα. Δηλαδή οι Βρετανοί θα πετάνε στον περιστερεώνα, μετά θα πετάνε από τον περιστερεώνα και εμείς θα περιμένουμε. πότε θα ε, μπορέσουν αυτοί που επιλέξαμε για να τους αντικαταστήσουν ε, αυτούς που αποχωρούν. Ο Μπάνξι, όπως ξέρετε, έκανε ένα ωραίο σχέδιο που φτιά, ε, εικονίζει το Westminster σαν να είναι γεμάτο με μαϊμούδες και ίσως να κάνει και άλλο ένα που θα κάνει το δικό μας σώμα γεμάτο με περιστέρια. Μια άλλη εικόνα. Φοβάμαι λοιπόν ότι με αυτή την απόφαση η πίεση για να υπάρξει διακομματική συμφωνία, όπως ανέφερε ο κύριος Καμάλ, θα εξαφανιστεί. Και τα δύο κόμματα μπορεί για άλλη μια φορά να επανέλθουν σε αυτό που κάνουν εδώ και μήνες, να περιμένουν να λήξει η προθεσμία. Και η απόδειξη είναι ότι η πρώτη απόφαση που πήρε, η πρώτη απόφαση που πήρε μετά από αυτή την τελευταία εξέλιξη το Βρετανικό Κοινοβούλιο ήταν να διακόψει για τις διακοπές του. Δεν περίμενα να ε, το πω αυτό, αλλά ίσως το μόνο που μπορεί να μας σώσει είναι ο Νάιτζολ Φαράτζ. Γιατί όπως θα ακούσετε, σήμερα ήδη κάνει προλογική εκστρατεία. Έχει δημιουργήσει ένα νέο κόμμα, το κόμμα για τον Brexit, για να προσπαθήσει να υπερκεράσει τους συντηρητικούς. Και τα δύο μεγάλα κόμματα, η συντηρητική και η εργατική, υπάρχει κίνδυνος να υποστούν τεράστια ήττα στις ε, ευρωεκλογές. Η συμβουλή μου λοιπόν προ αυτά τα δύο κόμματα είναι αν δεν είναι ανόητα κόμματα πρέπει να καταλήξουν συμφωνία τι επόμενε μέρε για να αποφευθεί αυτή η καταστροφή. Και κύριε Τάσκ, την επαύριο αυτή τη απόφαση είπατε κάτι το οποίο επαναλάβατε και τώρα πριν από λίγο. Είπατε ότι μπορεί να αποφύγουμε την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Και κοιτάξτε, και εγώ είμαι κατά τη αποχώρηση, αλλά δεν είναι δική μα απόφαση. Είναι απόφαση του Βρετανικού λαού. Φόβο μου λοιπόν είναι ότι αντί να σκοτώσουμε τον Brexit, η απόφαση μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο θανάτου για την Ευρώπη. Δηλαδή να βαλτώσουμε και πάλι για χρόνια. Όλη η ενέργειά μα να πηγαίνει σε διαπραγματεύσει με του Βρετανού ηγέτε. Όπω ο κύριο Κόρμπιν ή ο κύριο Τζόνσον. Οι οποίοι στην πραγματικότητα είναι κατά τη Ευρώπη. Τη συχαίνονται. Ενώ χρειαζόμαστε όλοι μα την ενέργεια για να μεταρρυθμίσουμε, για να ανεώσουμε την ε, ε, δική μα Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό Πρέπει και εσείς να εστιάσετε ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε αυτά. Και αυτού του είδους η προσέγγιση ήταν απούσα κατά τη γνώμη μου την περασμένη Τετάρτη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κυρία Τσίμερ, παρακαλώ, δύο λεπτά. Κυρίες και κύριοι, Υπάρχουν στιγμές νομίζω όπου οι αντιπαραθέσεις ε, για τις εκλογές πρέπει να σταματούν. Μας έδειξε, η χτεσινή για στο Παρίσι, πόσο ευάλωτος είναι ο κόσμος μας, πόσο εύθραυστη η Ευρώπη, ο πολιτισμός, η ιστορία και το μέλλον μας μαζί. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει πάντα να έχουμε υπόψη. Η Παναγία των Παρισίων είναι σύμβολο, σύμβολο της Ευρώπης, σύμβολο της Γαλλίας. Εγώ πριν από πολλά χρόνια Ανατολικογερμανίδα ξεκίνησα να μαθαίνω γαλλικά και ήξερα ότι θα μπορώ να έρθω να δω την Παναγία των Παρισίων. Είναι μεγάλο το σοκ λοιπόν για όλους μας εδώ, τους συναδέλφους. Και λέμε σε όλους τους Γάλλους ότι είμαστε στο πλευρό σας, αλλά ταυτόχρονα απαιτούμε να αναγνωριστεί πόσο ευαίσθητο, ευάλωτο είναι όλο αυτό αυτή η πολιτιστική κληρονομιά όπως και η Ευρώπη και με πόση προσοχή πρέπει να την αντιμετώπισουμε. Ούτε εγώ είμαι ικανοποιημένη από την έκβαση και τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής. Βρίσκω ότι είναι μοιραία απόφαση αυτή που ελήφθη γιατί ό,τι απόφαση και ληφθεί υπέρ ή κατά, επί έξι μήνες παρατείνεται αυτή η έκβαση και, σημαίνει και αυτό σημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βρίσκεται δεσμευμένο σε μια τέτοια ε, εξέλιξη επί ένα εξο, εξάμεινο. Δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Θα γίνουν οι εκλογές, θα περάσει η θερινή περίοδος, θα αρχίσουν οι ε, συγκροτήσεις ομάδων και κοινοβουλίου, θα είναι οι Βρετανοί μέσα ή έξω, θα έχουμε ένα ε, σχέδιο Α, ένα σχέδιο Β. Θα λέμε ότι έχουμε επιτροπές με μέλη τάδε και τάδε, πρόεδρος τάδε και δίνα, αλλά στην περίπτωση που θα υπάρχουν οι άλλοι, θα ε, υπάρχει διαφορετική σύνθεση ή και δύναμη των ομάδων. Έχετε σκεφτεί τι είναι αυτό με το οποίο μπορούμε να συνερπάσουμε τον πολίτη για την Ευρώπη σήμερα. Ήδη είναι τόσο δύσκολο όταν ξέρουμε ότι εκ των προτέρων βλέπει ένα τσίρκο ο πολίτης είναι δυνατόν να, μην, να δεσμεύεται το Κοινοβούλιο για, την επόμενη, για τους επόμενους μήνες και να μην είναι ξεκάθαρη κατάσταση για όλη τη θητεία. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ. Κυρία Σκοτκάτο, ένα μισή λεπτό. Πρόεδρε, έφτασε Πάσχα και είμαστε ακόμα εδώ. Χαίρομαι ιδιαίτερος και εγώ και τα εκατομμύρια των Βρετανών συμπολιτών μου. Χαίρομαι που μπορώ να ολοκληρώσω τη θητεία που μου εμπιστεύτηκαν οι ψηφοφόροι της Νοτιοανατολικής Αγγλίας και του Γιβραλτάρ πριν από πέντε χρόνια. Εμείς αυτό το εξάμεινο θα το αξιοποιήσουμε. Εμείς οι πράσινοι την προεκλογική εκστρατεία θα την αξιοποιήσουμε για να προβάλλουμε τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα είμαστε μια από τις πιο ισχυρές δυνάμεις και θα υπερασπιστούμε στην Ευρώπη μια, μια πιο πράσινη Ευρώπη, μια πιο δημοκρατική και πιο ισχυρή Ευρώπη και ευχαριστώ τον πρόεδρο Τούσκ που μας έδωσε αυτό το περιθώριο να πάρουμε μια ανάσα και να ξανασχεδιάσουμε το μέλλον μας. Ποτέ δεν ήταν ευχερής η οικοδόμηση της Ευρώπης. Ο κύριος Τούσκ παρέπεμψε στο ιστορικό και τους ιδρυτές της Ευρώπης οι οποίοι έκαναν προσπάθειες για να συμπεριλάβουν και να κρατήσουν στην Ευρώπη αυτούς που είχαν και στο εσωτερικό τους, στο εσωτερικό της χώρας τους δυσκολίες. Εγώ ω πράσινη πάντοτε ήμουν σκληρή επικρίτρια του Brexit, αλλά πρέπει να είμαστε σκληροί επικριτέ και στα αίτια που οδήγησαν στο Brexit. Δηλαδή την ιδέα που έχει ο πολίτη ότι είναι αδύναμο, ότι έχει απομακρυνθεί, ότι δεν έχει κανένα λόγο στην Ευρώπη. Και αυτό οδήγησε στο αποτέλεσμα του δημοψηφίσματο του 2016. Για εκείνου λοιπόν του φίλου οι οποίοι ήταν υπέρ τη παραμονή του Ηνωμένου Βασιλείου, το μήνυμα ήταν, είναι α αξιοποιήσουμε αυτό που υπάρχει, ας προβάλλουμε τα καλά της Ευρώπης, ας καταρρύψουμε τις ειρήνες των ακροδεξιών. Πρέπει με τις επόμενες εκλογές να κερδίσουμε την ψήφο του πολίτη, να πείσουμε τον πολίτη, τον συμπολίτη μας ότι το καλύτερο μέλλον για το Ηνωμένο Βασίλειο είναι να παραμείνει κομμάτι αυτής της ευρωπαϊκής οικογένειας. Mr. Farage, five minutes. Thank you. Good morning. Well, I have tried for 20 years Κοιτάξτε, εδώ και 20 χρόνια προσπαθώ να φύγω από εδώ πέρα. Και νόμιζα ότι είχα πετύχει. Αλλά δεν είχα καταλάβει τι θα έκανε η πολιτική τάξη του Ηνωμένου Βασιλείου. Και κοιτάξτε, το μήνυμά μου είναι θα ξανάρθω. Πολλοί από εμά θα ξανάρθουν. Γιατί ο κύριο Φαρχόφστατ έχει δίκιο. Ναι, ναι, το είπα. Ναι, ήμουν ο πρώτο που το είπα αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Το κόμμα του Brexit θα σκίσει σε αυτέ τι εκλογέ. Και μόνο ένα τρόπο είναι να το σταματήσετε. Είναι το κόμμα τη κυρία Μέη και η αντιπολίτευση του κ. Κόρμπιν να συμφωνήσουν και να συμφωνήσουν σε μια μόνιμη τελεωνική ένωση και στην ουσία ε, να είναι και μέλη τη ενιαία αγορά. Αν γίνει αυτό, το κόμμα του Brexit δεν θα κερδίσει τι ευρωεκλογέ. Θα κερδίσει τι εθνικέ εκλογέ. Γιατί η προδοσία θα είναι τόσο ολοκληρωμένη και καταφανής. Δεν νομίζω γι' αυτό ότι θα συμβεί αυτό. 15 χρόνια που είμαι πρόεδρος ε, ε, με άλλους ή μόνος μου ενός πολιτικού κόμματος, έχω συμμετέχει, συμμετάσχει σε πολλές συναντήσεις κορυφής και έχω δει πολλές συγκρούσεις μεταξύ κρατών και των ευρωπαϊκών ε, θεσμών, η Αυστρία, η Ιρλανδία, η Ουγγαρία ή η Ελλάδα. Και υπάρχει ένας χρυσός κανόνας. Πάντα. Είναι ότι κερδίζει οι Βρυξέλλες. Η ισχύ των Βρυξελών τα καταφέρνει πάντα να κερδίσει. Αλλά ποτέ δεν πήγα σε συνάντηση κορυφή όπω την προηγούμενη εβδομάδα. Όπου για δεύτερη φορά σε δύο εβδομάδε μια Βρετανίδα πρωθυπουργό έρχεται και ζητιανεύει, ζητιανεύει. Ε, παρακαλά για μια παράταση του άρθρου 50. Ήταν ξεφτύλα. Όχι μόνο να είναι κανεί στι Βρυξέλλε. Ξεφτύλα, ταπεινωτικό για τη χώρα μα. Την θέση στον κόσμο. Ξέρετε, έχουμε την κοινοπολιτεία, το οι Ηνωμένε Πολιτείε. Υπάρχουν πολλέ χώρε που μα γουστάρουν. Θεωρούν ότι είμαστε ακόμα ένα μεγάλο έθνο. Και όμω έχουμε πέσει τόσο χαμηλά. Η Πρωθυπουργό που μα υποσχέθηκε ότι θα φύγουμε στι 29 Μαρτίου είπε ε, μπορεί να φύγουμε στις 12 Απριλίου. Θα φύγουμε οπωσδήποτε στις 30 Ιουνίου. Και τώρα τι μας λέει. Θα φύγουμε 31 Οκτωβρίου. Θα είναι Halloween δηλαδή. Ή γλυκό ή φάρσα. Ε, ελπίζω, ελπίζω να αποχωρήσουμε τελικά. Αλλά αν το αφήσουμε σε αυτή την άθλια πρωθυπουργό αν αφήσουμε του ε, πολιτικού μα στο κοινοβούλιο να χειριστούν το θέμα, δεν θα συμβεί ούτε αυτό. Στο παρελθόν ξέρω ότι πάντα επέκρινα τη δύναμη χωρίς λογοδοσία των ε, κυρίων ε, γραφειοκρατών των Βρυξελών. Αλλά πρέπει αυτή τη φορά να πω ότι για αυτά τα χάλια δεν φταίτε εσεί. Από την αρχή είχατε σαφή θέση. Αυτά τα χάλια είναι ευθύνη των δύο μεγάλων Βρετανικών κομμάτων που και τα δύο μας υποσχέθηκαν στα προεκλογικά τους προγράμματα ότι θα υπάρξει Brexit που δέχθηκαν να πυροδοτηθεί το άρθρο 50 που είπαν ότι θα φύγουμε με συμφωνία χωρίς. Μας πρόδωσαν, αυτοί μας πρόδωσαν. Και συμφωνώ την, ε, με τη θλίψη που εξέφρασαν και οι άλλοι για την καταστροφή χθε της Νορνταν. Κάτι τόσο όμορφο καταστράφηκε αλλά ε, χάνεται και κάτι άλλο πολύ ζωτικό για το Ηνωμένο Βασίλειο. Και νομίζω ότι χθε ε, οι νεκρολογίε του Times το έλεγαν. Πολύ σωστά. Ε, η νεκρολογία έλεγε ότι η δημοκρατία του Ηνωμένου Βασιλείου 312 ετών πέθανε στις 29 Μαΐου. Πέθανε ίσχα στον ύπνο της στις 11 το απόγευμα στις 29 Μαρτίου 2019. Αιτία θανάτου, δολοφονία και οι ένοχοι ακόμη δεν έχουν εντοπιστεί. Η δημοκρατία ε, ήταν ε, κάτι το οποίο στήριζε ε, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις δημοκρατικές αποφάσεις. Θα μας λείψει ο Θεός να μας βοηθήσει. Αυτό που θα γίνει στις 23 Μαΐου δεν έχει να κάνει μόνο με τον Brexit και την αποχώρησή μας από την Ένωση. Είναι για το τι είδους χώρα είμαστε. Έχουμε την παλιότερη κοινοβουλευτική παράδοση στον κόσμο. Τη μητέρα των κοινοβουλίων. Αγωνιστήκαμε και δώσαμε πολλά για αυτή την αρχή τη δημοκρατία ενό εθνικού κράτου, όχι μόνο για εμά, αλλά για του φίλου μα στην Ευρώπη. Και ορισμένοι εδώ, στη χώρα μου μάλλον καλύτερα, είναι απογοητευμένοι. Αλλά άλλοι είναι τρομερά αγανακτισμένοι. Δεν βάζουν κίτρινα γυλαίκα εκείνοι. Αλλά λένε, χρειαζόμαστε μια ειρηνική πολιτική επανάσταση στη χώρα μου. Πρέπει να εξαφανιστούν τα δύο αυτά κόμματα τα οποία μας πρόδωσαν. Και νομίζω ότι όλοι σας θα εκπλαγείτε ιδιαίτερα από αυτά που θα συμβούν στις 23 Μαΐου. Θα είναι μια καινούργια αρχή για τη Βρετανική Δημοκρατία και πραγματικά τη χρειαζόμαστε. Συνάδελφοι, λέει πρόεδρος, έλαβα κάποια αιτήματα για μπλε κάρτα. Αλλά επειδή Υπάρχει ήδη προηγούμενο, δεν υπάρχουν μπλε κάρτε κατά τη διάρκεια τη συζήτηση των ηγετών. Και τώρα ο κύριο Μπάτεν, τρία λεπτά. Όλα αυτά δεν θα έπρεπε ποτέ να συμβαίνουν. Αν είχε τιμηθεί η απόφαση του δημοψηφίσματος το 2016 και η Βρετανία είχε φύγει εδώ και πολύ καιρό. Ωστόσο, η δημοκρατική απόφαση 17,4 εκατομμυρίων ανθρώπων η θελημένα προδίδεται. Οι ευρωεκλογέ του Μαΐου αναπόφευκτα θα είναι μια επανάληψη του δημοψηφίσματος. Όποιο, ό,τι και αν πούνε τα πολιτικά κόμματα, η επιλογή των ψηφοφόρων θα είναι στην ουσία επί του αν θα μείνουμε ή θα φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπέρ του να μείνουμε θα πρέπει να ψηφίσουν τους ε, φιλελεύθερους δημοκράτες. Είναι το κόμμα του παραμένουμε. Ενώ αυτοί που θέλουν να φύγουν θα πρέπει να, ψηφίσουν το κόμμα της ε, ανεξαρτησίας. Το UKIP είναι ε, το κόμμα που θα προχωρήσει στην έξοδο. Οι υπόλοιποι δεν ξέρουν ούτε καν τι θέση έχουν για αυτό το θέμα. Η πολιτική του UKIP είναι σαφής ε, και ξεκάθαρη. Είναι της μονομερούς και ανεφόρων εξόδου. Αυτέ όμω οι εκλογέ θα διχάσουν τον κόσμο σε δύο διακριτές ομάδε, όχι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η μια ομάδα θα είναι αυτή που συγκατατίθεται να του κυβερνεί να μια ξένη δύναμη, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δεύτερη ομάδα θα είναι αυτή που επιλέγουν να επαναστατήσουν ενάντια σε περαιτέρω ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και υπέρ τη επιστροφή των δημοκρατικών ε, αξουσιών στα κράτη-έθνη. Η μια ομάδα θα αγωνίζεται για την ελευθερία και την ανεξαρτησία, η άλλη ομάδα θα ψηφίσει υπέρ της υποδούλωσης και της υποταγής. Κάτι για το οποίο ε, ε, πρέπει να είμαστε βέβαιοι είναι ότι οι ευρωσκεπτικιστέ, οι ευρωβουλευτέ θα επανέλθουν πολύ ε, άριθμοι, πολύ άριθμοι και οι ψηφοφόροι του θα ψηφίσουν υπέρ τη επιστροφή στη δημοκρατική λογοδοσία, στο τέλο των μέτρων λιτότητα και στην διαχείριση των οικονομιών προ το συμφέρον του και το όφελό του θα ψηφίσουν υπέρ τη πάυση τη μαζική και ανεξέλεγκτη μετανάστευση. Θα ψηφίσουν υπέρ κομμάτων που θέλουν να διατηρήσουν τον πολιτισμό του και την κουλτούρα του. Και θα το, UKIP θα, είναι η ψήφο, η λαϊκή ψήφο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε την ψήφο υπέρ του παραμένουμε ή του υπέρ του φεύγουμε οι ε, εκλογέ τι οποίε παρότρινε το UKIP έφεραν το δημοψήφισμα και το UKIP θα εξακολουθήσει τον αγώνα ώστε να γίνει πραγματικότητα το Brexit. Στι 31 Μαου οι βουλευτέ του UKIP θα συνεχίσουν τον πολιτικό αγώνα ώστε να απελευθερωθεί το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία ψήφο υπέρ του UKIP στις 31 Μαου θα στείλει σαφέ μήνυμα στην κυβέρνηση να φύγουμε και από το ΠΟΕ άμεσα. Το UKIP δεν είναι μόνο μια εκστρατεία υπέρ του Brexit. Θέλουμε αυτό να γίνει πραγματικότητα. Μια ψήφο στο UKIP σημαίνει πάντα αποχώρηση από την, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι Βρετανοί θα πρέπει να ψηφίσουν υπέρ του UKIP στις 31 Μαΐου. Ο κύριος και ένα λεπτό παρακαλώ. Μια εγγεγραμμένος. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Το θέμα του καθεδρικού ναού της Πανηγίας των Παρισιών στις Φλόγες ήταν ε, εικόνα τραγική. Όλοι βέβαια, υπόθηκε νωρίτερα, πρέπει να αντιληφθούμε ότι έρχεται η στιγμή που πρέπει να λάβουμε τις δύσκολες αποφάσεις. Καλωσορίζω την απόφαση του Συμβουλίου για την παράταση της προθεσμίας του Brexit. Απεφεύχθη το μοιραίο, η σύγκρουση. Μόνο αυτοί που, μόνο αυτοί που είναι κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και του Ηνωμένου Βασιλείου ε, είναι δυσαρεστημένοι. Και βέβαια ο κύριος Φαράζος δεν με ξάφνιασε. Με ξάφνιασε όμως ο κύριος Φερχόφστατ, που φαίνεται φεντεραλιστής όν, να κάνει τη δουλειά των λαϊκιστών. Δηλαδή να λέει ότι πρέπει να φύγει το Ηνωμένο Βασίλειο. Όχι, δεν είναι αυτή η λύση. Χρειάζεται πραγματισμό, ρεαλισμό, συνεργασία. Ελπίζω με την προσεχή ε, περίοδο τη βουλευτική να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε τον δρόμο αυτό. κύριο Μπροκ, ένα λεπτό και 30 δεύτερα. Πρόεδρε, Πρόεδρε του Συμβουλίου, Πρόεδρε τη Επιτροπή, αγαπητοί συνάδελφοι, θα έχουμε νέα κατάσταση, νέε συνθήκε τον Οκτώβριο ή θα ξαναζούμε την ίδια κατάσταση με αυτή που έχουμε σήμερα γιατί θα έχει λυθεί το ζήτημα. Ελπίζω να βρούνε μια λύση ο Κόρμπιν και η Μέη. Να πιέσουν το, τη Βουλή των Κοινοτήτων να βρούνε μια επικοδομητική λύση είτε για να μείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε για να αποχωρήσουν πάντως όχι με ε, μεσοβέζικες λύσεις, λύσεις και πρέπει εμείς να κοιτάξουμε πλέον να ασχοληθούμε με τα μεγάλα προβλήματα που μας περιμένουν στο μέλλον, τα ζητήματα της μετανάστευσης, των πολέμων των εμπορικών συναλλαγών, των, ε, της ασφάλειας τα εξωτερικά σύνορα, σύνορα της κλιματικής αλλαγής και πολλά άλλα. Πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η μόνη δύναμη με την οποία μπορούμε όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε τις, μεγά, τις μεγάλες απειλές των Τραμπ και των του Πούτιν του κόσμου και να σώσουμε έτσι την Ευρώπη και να τις επιτρέψουμε επιτρέψουμε να προοδεύσει. Έτσι πρέπει να συνεχίσουμε ως μια μεγάλη δύναμη και να μην επιτρέψουμε το διχασμό που φέρνει ο λαϊκισμός. Έτσι λοιπόν με την Ευρώπη αυτή, την Ευρώπη της αλληλεγγύης, της ειρήνης, της ελευθερίας, της ανθρωπιάς, της ε, επιτυχίας της Ευρώπης αυτής ε, η οποία έχει εξασφαλίσει τόσα πολλά για όλο τον κόσμο, για όλους τους πολίτες. Ύστερα από 39 χρόνια η τελευταία μου ομιλία είναι η σημερινή και με αυτήν θέλω να σημειώσω ότι η Ευρώπη στέφθη με επιτυχία στην ιστορία της ε, ανθρωπότητας. Σε νέα κράτη ήμασταν όταν εγώ πρωτοέγινα βουλευτής. Ε, και δεν λειτουργούσε ακόμα καλά-καλά η Τελωνιακή Ένωση. Τώρα έχουμε φτάσει στα 28 κράτη-μέλη και πρέπει αυτή την ένωση να την τιμήσουμε και να ε, εξηγήσουμε και στον πολίτη, στον ψηφοφόρο γιατί είναι τόσο σημαντική. Μπορεί να μην είναι μόνο ένα ωραίο ε, κτίριο ή ε, ναός η Παναγία των Παρισίων είναι πολιτιστική κληρονομιά πάνω απ' όλα, όχι μόνο της Γαλλίας αλλά όλης της Ευρώπης και όλου του κόσμου. Και θυμάμαι τη στιγμή εκείνη που Κάναμε την επιμνημόσυνο δέηση για τον Helmut ε, με τον Helmut Kohl για τον François Μιτερό. Είναι η στιγμή η οποία δεν μπορεί να ξεχάσει κανείς, μια στιγμή ενότητας και ήρθε ο François Μιτερό εδώ στο Κοινοβούλιο για να πει λέει συγκινημένο ο ομιλητή, ότι ο, ο εθνικισμό ε, στο δυναμεί με πόλεμο. Αυτά τα λόγια δεν πρέπει να τα ξεχάσουμε ποτέ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπροκ. Είναι τελευταία σας ομιλία στο σώμα μας. Υπηρετήσατε ιδιαίτερα καλά το σώμα και ελπίζω να μην ξεχάσετε τελώς την ευρωπαϊκή πολιτική. Τώρα θα την αντιμετωπίζετε από άλλη οπτική γωνία. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι το σώμα απέτυσε φόρο τιμής με το χειροκρότημά του σε εσά. It's one of those emotional ε, ε, κύριε Μπρόκ, ε, υπάρχει πολύ συγκινησιακή φόρτιση ε, σήμερα το πρωί και νομίζω ότι διαπιστώνετε πόσο εκτιμούν οι συνάδελφοί σα. Ο κύριο Κόρμπετ, τώρα για δύο λεπτά, ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να συμφωνήσω με όσου αναφέρθηκαν στην τραγωδία του Νότρο Ντάμ και ιδιαίτερα αυτά που είπατε εσεί, ότι και εμεί μεριζόμεθα τον πόνο του γαλλικού λαού. Είπατε ότι δεν μα συνδέουν απλώ συνθήκες και κείμενα. Αυτό ισχύει. Και γι' αυτό ε, σκανδαλίστηκα όταν τη στιγμή που το λέγατε αυτό ο κύριος Φαράτζ, ο οποίος έχει ήδη φύγει ως συνήθως, φώναξε βλακίες. Αυτό νομίζω ότι αποδεικνύει τη στάση πολλών από την άλλη πλευρά. Αλλά είναι η φωνή του παρελθόντος. Ο Βρετανικός Λόγος αρχίζει να καταλαβαίνει τι ψέματα του λένε εδώ και χρόνια για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρχίζουν να βλέπουν τα ψέματα που τις είπατε για τον Brexit. Μας είπατε ότι θα ήταν πολύ εύκολο. Ε, είναι αρκετά περίπλοκο, ε. Μας είπατε ότι θα εξοικονομούσαμε πολλά χρήματα για το σύστημα υγεία μας. Τελικά θα μας κοστίσει μια περιουσία. Μας είπατε ότι θα έχουμε έτοιμες νέες εμπορικές συμφωνίες με χώρες παντού στον κόσμο για να αντικαταστήσουν ε, το εμπόριο που θα χάσουμε από την Ευρώπη. Χάνουμε όλες τις ε, συμφωνίες που έχουμε μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν υπάρξει Brexit. Ο Βρετανικός λαός αρχίζει να αντιλαμβάνεται τι του είπαν. Και γι' αυτό φοβούνται τόσο πολύ το να γίνει ένα νέο δημοψήφισμα. Γιατί ξέρουν ποια θα ήταν η απάντηση αν υπήρχε νέο δημοψήφισμα. Γι' αυτό οι συντηρητικοί δεν θέλουν να γίνουν ευρωεκλογέ. Γιατί ξέρουν ότι θα συντριβούν σε αυτέ τι εκλογέ. Και εκπλήσω με λιγάκι που ο κύριο Φερχόφστατ και ορισμένοι άλλοι εδώ στο σώμα μα, εδώ φοβούνται αυτέ τι εκλογέ. Γιατί φοβάστε, δεν υπάρχει λόγο. Η πλειονότητα των ευρωβουλευτών που θα επιστρέψουν δεν θα είναι του φυράματος των απέναντι. Και, εν πάση περιπτώσει, εν περιπτώσει, το Brexit, η αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ενός μέλους για πρώτη φορά, οι επιπτώσεις αυτής της απόφασης είναι πολύ πιο σημαντικές από το συσχετισμό δυνάμεων των πολιτικών ομάδων δείτε τα πράγματα στο σωστό πλαίσιο. Αυτή η παράταση πρέπει να αξιοποιηθεί όπως σωστά είπε ο κ. Τούσκ. Εντάξει, δεν έχω και πολλές ε, μεγάλες προσδοκίες για ε, τη συζήτηση μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων. Γιατί η κυρία Μέρη μπορεί να αλλάξει θέση χωρί να αντιμετωπίσει ανταρσία από το κόμμα τη, αλλά μα δίνει μια ευκαιρία να επανέλθουμε στο λαό και να σταματήσει αυτό το άθλιο χάλι στο οποίο έχουμε καταλήξει. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Νίκολσον, ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να συμφωνήσω με την έκφραση παράσταση προς τον γαλλικό λαό σήμερα το πρωί. Όλοι ε, αισθανόμαστε τι αισθάνονται. Οι τελευταίες εξελίξεις, η περαιτέρω παράταση της αβεβαιότητας, αναβολητικότητα δηλαδή, είναι αυτό που συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, η παράταση αυτή μα δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε το πραγματικό πρόβλημα. Αλλά δεν θα εκπλαγείτε κύριε Μπαρνιέ γιατί εγώ θεωρώ ότι το πρόβλημα αυτό είναι το backstop. Δεν είχα αλλάξει άποψη από αυτού. Το backstop έχει δυσχεράνει τι διαπραγματεύσει από την αρχή και θα συνεχίσει να το κάνει όσο εμένετε στη θέση σα. Πρέπει να σα πω ότι η παράταση μέχρι τον Οκτώβριο δεν νομίζω ότι θα καταλήξει σε συμφωνία. Θεωρώ ότι θα χρειαστεί μια νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ένα νέο Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να αλλάξουν απόψει. Θα πρέπει να δοθεί μια ε, νέα ευκαιρία για να απαντήσουμε αυτό το πρόβλημα. Κοιτάξτε, εάν είναι κανεί μέλο μια λέσχη, πρέπει να είναι πλήρε μέλο. Δεν μπορεί να είσαι μισό μέσα και μισό έξω. Και αυτό είναι το πρόβλημα με το Ηνωμένο Βασίλειο. Αν μου επιτρέπετε. Έχει φύγει ο κύριο Μπροκ, αλλά παρόλα αυτά θα είναι και η δική μου τελευταία ομιλία σε αυτό το σώμα μετά από 30 χρόνια. Και θέλω να αξιοποιήσω την ευκαιρία για να σας πω ότι ήταν μεγάλη μου τιμή αλλά και χαρά να εκπροσωπήσω το λαό της Βόρειας Ιρλανδίας σε αυτό το σώμα για 30 χρόνια. Τα πήγαμε καλά ορισμένε φορές και, μερικέ, και μερικές φορές ήταν ε, πολύ άσχημες οι καταστάσεις που αντιμετωπίσαμε όταν είχαμε και τρομοκρατικές επιθέσεις όπως εδώ. Και περάσαμε όλοι μέσα από αυτά. Αλλά στο σώμα αυτό ακούσαμε τον Ζακ Ντελόρ που εξέφρασε την αλληλεγγύη του με τον πληθυσμό της ε, Βόρειας Ιρλανδίας και όταν εγώ, ο Ιαν Πέισλι και ο Τζον Χιούμ πήγαμε να τον δούμε, μας ρώτησε τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη για σας και η Ευρώπη βοήθησε, έδωσε πάνω από δύο δις που βοήθησαν πολλούς ανθρώπους παντού στη Βόρεια Όπως είπα και εγώ, λοιπόν, σας ε, αποχαιρετώ. Ελπίζω να συνεισέφερα εγώ πέρασα καλέ καταστάσει. Ελπίζω να προσώπησα σωστά το λαό μου, γιατί είναι ένα περήφανο λαό, είναι ένα καταπληκτικό λαό, ο λαό τη Βόρεια Ιρλανδία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Νίκολσον. Και επειδή έχουμε δουλέψει μαζί, στην Επιτροπή Γεωργίας πρέπει να πω ότι όντως είχατε πολύ επικοδομητική στάση εκπροσωπώντας τα συμφέροντα των εκλογέων εδώ και 30 χρόνια. Σε ευχόμαστε ότι καλύτερο. Νομίζαμε ότι οι προηγούμενοι ομιλίες θα ήταν τελευταία, αλλά τελικά είχατε μια δυνατότητα ακόμη. Συγγνώμη που ε, δεν τηρώ το χρόνο τώρα. Και τώρα κύριε Άντερσον για λεφτό. Τίποτα δεν έχει αλλάξει. Το Λονδίνο παραβιάζει επιλεκτικά τις συμφωνίες Μεγάλης Παρασκευής. Το Δουβλίνο μας παραμελεί εμάς το Βορρά. Άλλοι έξι μήνες αβεβαιότητας διότι οι Βρετανοί αναβάλουν αυτά τα οποία συμφώνησαν ότι πρέπει να εφαρμόσουν το Δεκέμβριο του 2017. Το Brexit τους ε, αφαιρεί τα δικαιώματα του, του λαού συμπεριλαμβανόμενο και το δικαιώματο ψήφου, κάτι που ήταν ε, στην καρδιά του κινήματο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τα πολιτικά δικαιώματα. Αντιμετωπίζουμε λοιπόν εκλογέ που η συντηρητική και το DUP δεν ήθελε και που τα δύο κόμματα τη ε, Νότια Ιρλανδία δεν ήθελαν να ψηφίσει ο Βορρά για αυτά. Α στείλουμε ένα σαφέ μήνυμα στο Λονδίνο, το Δουβλίνο και τι Βρυξέλλε. Α ε, επικρίνουμε το χάλι του Brexit αυτό τον πολιτικό μανδαλισμό. Όλοι οι ψηφοφόροι στην Ιρλανδία, εκλέγοντα ευρωβουλευτέ του Sinn Féin, μπορούν να κάνουν ένα βήμα προς την Ιρλανδική ενότητα που θα είναι ο δημοκρατικός τρόπος για να βγούμε από το Brexit. Θα είναι μια σωστή λογική απόφαση για να επιτύχουμε την Ιρλανδική ενότητα. Σας ευχαριστώ όλους. Έχει ζητηθεί μπλε κάρτα. Κύριε Κέλλη. Παρακαλώ. Κύριε Άντερσον, εσείς δέχεστε να σας διατυπώσει την ερώτηση ο κύριος Σκέλη. Κύριε Σκέλη, ξέρετε ότι δεν συνηθίζω να ρωτάω με μπλε κάρτα του συναδέλφου. Είναι η δεύτερη μου τα δέκα χρόνια που είμαι εδώ. Αλλά όταν μας λέει η κυρία Άντερσον ότι έχει καταληφθεί η υπόθεση της Βόρειας Ιρλανδίας και όταν ξέρουμε ότι με τον backstop... Ένα λεπτό, ε, λέει η Πρόεδρος, κάντε την ερώτηση. Ναι, όταν όμως ε, δεν έρχονται να συμμετάσχουν σε κανένα κοινοβούλιο ή συνέλευση τα μέλη του κόμματός της. Μα βλέπετε ότι εγώ είμαι εδώ, κύριε Κέλλη. Το Σινφέιν ξεκάθαρα τοποθετήθηκε σε σχέση με την απόφαση της ε, Ιρλανδικής κυβέρνησης, η οποία είναι η μόνη η οποία στερεί το δικαίωμα της συμμετοχής στις ευρωεκλογές από τους υπηκόους της όταν δεν κατοικούν μέσα στην επικράτεια της Ιρλανδικής Δημοκρατίας. Το ξέρεις πολύ καλά, Τζον, Σον, όταν με τον Τζον Χιούμ πήγαν η μητέρα μου και ο πατέρας μου και όλοι οι συγγενεί μου στο Λονδίνο να αγωνιστούν με τα συλλαλητήρια ζητώντας ψήφο ισότιμη, δεν είχαν την εκπροσώπηση, δεν είχαν τη δυνατότητα. Ευχαριστώ πολύ, λέει η πρόεδρος. Τέλειωσε ο χρόνο σας. Κύριε Σμιθ, για ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ε, βεβαίως και είναι κάπως υπερβολικές όλες αυτές ε, οι δηλώσεις περί αποτυχίας και κατάρρευσης, αλλά θα ήθελα να πω, Πρόεδρε Τούσκ, ε, όπως, λέει και ο, όπως έλεγε ο Τζον Λένον, μπορεί να είσαι ονειροπόλος, αλλά δεν είσαι ο μόνος. You're a dreamer, but you're not the only one. Ευχαριστώ λοιπόν για τις προσπάθειές σας, κύριε Τούσκ, και το χρόνο που αφιερώσατε για τη διέξοδο. Ε, ωστόσο, και εν των ευρωεκλογών, θέλω ένα μήνυμα να αποστείλω. Να αποκομίσουμε όλοι το δίδαγμα του Brexit, να το μάθουμε το μάθημα αυτό, γιατί το Brexit ε, καραδοκεί σε κάθε χώρα. Οι λαϊκιστές είναι επικίνδυνοι παντού και πρέπει να αποστείλουμε και θεωρώ ε, παρατηρητές στις εκλογές γιατί δεν θα είναι απαραίτητα καθαρή η εκλογική αναμέτρηση. Θα ήθελα να βεβαιωθούμε ότι θα γίνει γνήσια εκλογική αναμέτρηση και επίσης ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι μπορεί να προσπαθήσουν να εμποδίσουν την ανάδειξη καθαρού αποτελεσμού από τις εκλογές και αν το ξανακάνουν το κόμμα μου στην Σκοτία είναι έτοιμο για να γυρίσει στην Ευρώπη και θέλουμε να στηριζόμαστε σε εσά όπως μπορείτε και εσείς να στηρίζετε σε εμά. Η κυρία Γκέρλινγκ για ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εδώ παρισταμένους για την υπομονή, αλλά και την ηγετική στάση που επέδειξαν σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, κύριε Τούσκ, ιδιαίτερος προς εσάς πρέπει να ε, ε, πω ευχαριστώ με όλα ε, στις επιστολές, τα γράμματα που έχω λάβει που μου λένε πηγαίνετε να βρείτε τον Τούσκ, η μου, να του σφίξετε το χέρι, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις προσπάθειές του. Έχετε αναλάβει μια ευθύνη βαριά, μια ευθύνη να αντιμετωπίσετε την εκδοχή της ε, εξόδου του Ρωμανού Βασιλείου χωρίς συμφωνία και αυτό ήταν μια βαριά ευθύνη για να αντιμετωπίσετε τα λάθη των συντηρητικών που έκαναν προχειροδουλειά και προκυρήσοντας ένα δημοψήφισμα για το οποίο δεν ήταν έτοιμοι. Η δουλειά του κυρίου Μπαρνιέ, του κυρίου Τούσκ, του κυρίου Γιουνκέρ πολιτικών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ήταν αυτοί που μας επιτρέπουν να συμμετάσχουμε στις 23 Μαΐου που διεξάγονται οι ευρωεκλογές στη Βρετανία και τους ευχαριστούμε γι' αυτό διατηρούμε την ελπίδα να μείνουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην ε, Ηνωμένη Ευρώπη και είναι γενναίοι εκείνοι οι οποίοι βάζουν το μέλλον της χώρας μπροστά από τα μικροκομματικά συμφέροντα. Ήρθε η ώρα να ζητήσουμε να γίνει δημοψήφισμα το Σεπτέμβριο, έτσι ώστε έως τις 31 Οκτωβρίου να έχει ληφθεί απόφαση ότι θα παραμείνουμε, ότι θα επικρατήσει το Remain. Ευχαριστώ, κύριος Ντάνς, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα ε, στα γαλλικά να εκφράσω εκ μέρους του λαού της Ιρλανδίας ε, τη συμπόνια μας προς το λαό του Παρισιού για την καταστροφή της Πανηγίας των Παρισίων. Θα την ξαναχτίσουμε όλοι μαζί. Θέλω να τιμήσω και το θάρρος των πυροσβεστών. Συνάδελφοι, το Brexit είναι μια διαδικασία εν την οποία αρνούνται αυτοί που κάθονται απέναντί μου, αρνούνται να κοιτάξουν ότι κάθε επιλογή που έχει μέσα της ένα Brexit, μια έξοδο, έχει αρνητικές συνέπειες τους. Είναι πολύ πιο εύκολο λοιπόν να κάθονται και να λένε «Α, μας προδώσατε» χωρίς όμως να πράττουν τίποτα, γιατί το Brexit δεν μπορεί να υλοποιηθεί όπως το υποσχέθηκαν. Ελπίζω να μπορέσουμε να κάνουμε νέες εκλογές ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο, ώστε να δοθεί στο λαό η επιλογή να καταρρύψει όλους αυτούς που μιλούν για τα μονάχα Όλοι εμεί που είμαστε διατεθειμένοι από αυτήν εδώ την πλευρά να σταθούμε ε, στο πλευρό των Ευρωπαίων συμπολιτών μα και να χτίσουμε μαζί ένα κοινό μέλλον, είμαστε έτοιμοι να το πράξουμε. Σα ευχαριστώ. Κύριε Χένκελ, ένα λεπτό. Πρώτη φορά πήγαμε το ποδήλατο από το Λουξεμβούργο μέσω Βελγίου στο Παρίσι, ποδηλάτης, για να επισκεφθώ την ε, Παναγία των Παρισίων και χτες την είδα να φλέγεται και δάκρυσα. Κυρίες και κύριοι, είπατε κύριε Τούσκ ότι συμπονείτε το Παρίσι γιατί, είδατε, γιατί ξέρετε πως είχε καταστραφεί το Γκάνσκ. Θα σας μιλήσω εγώ για την ε, ε, Παναγία της Δρέσδης που χτίστηκε με την συνδρομή των Βρετανών των χτιστών που ήρθαν από το Κόβεντρι. Και θα πω ότι πρέπει να γίνει κοινό εγχείρημα για να ξαναχτιστεί η μεγάλη η Παναγία των Παρισιών, ο καθεδρικός ναός του Παρισιού. Πρέπει να είναι ένα κοινό εγχείρημα ευρωπαϊκό. Κύριε Τούσκ, είπατε επίσης ότι θα πρέπει και τα 28 κράτη να συμμετάσχουν. Την απάντηση πρέπει να τη δώσει το Λονδίνο βέβαια πια. Γιατί άκουσα και εσείς τι είπατε και ο κύριος Γιούνκερ. Αλλά κάτι πρέπει να πράξετε για να λάβετε τη σωστή απάντηση από το Λονδίνο. Αυτό πρέπει να πράξετε είναι να εξασφαλίσετε πως η Βρετανία θα παραμείνει και θα είναι μέλον, μέλος της προσπάθειας ανοικοδόμησης από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης της Παναγίας των Παρισίων για να μπορέσει να παραμείνει μέλος της ε, Ενωμένης Ευρώπης, του Ρωμένο Βασίλειο. Κυρία Χιούμπνερ, για ένα λεπτό. Eh, eh, Ευχαριστώ. Πρόεδρε, Πρόεδρε συνάδελφοι. Για τους Ευρωπαίους ηγέτες η νέα προθεσμία για τον Brexit ήταν δύσκολη απόφαση. Ε, τώρα η Βρετανική πλευρά θα πρέπει να χρησιμοποιήσει με επικοδημητικό τρόπο αυτό τον περαιτέρω χρόνο και σίγουρα δεν βασιζόμαστε στον κύριο Φαράζ. Είναι απογοητευτικό ότι την τελευταία εβδομάδα ακούσαμε σχόλια και είδαμε tweets ε, αντιευρωπαίων πολιτικών για το πώς θα σαμποτάρουν τη δουλειά μας στους επόμενους μήνες. Αυτή η πολιτική πρέπει να καταλάβουν ότι δεν πρόκειται να τους το επιτρέψουμε, θα προστατεύσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους πολίτες της. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξακολουθήσει να αποτελεί την πηγή της σταθερότητας για, σε αυτήν την παράλογη διαδικασία του Brexit. Δυστυχώς από την Βρετανική πλευρά δεν υπάρχουν μηνύματα, δεν υπάρχουν δείγματα ότι το μια συμφωνία για τον Brexit ε, θα επιτευχθεί. Το προβληματικό πρόβλημα δεν είναι το backstop, είναι το μέλλον. Και ίσως μια λύση να βρεθεί. Αυτό που χρειάζεται στη βρετανική πολιτική είναι το να οριστεί, να αποφασίσουν τι πραγματικά θα επιθυμούν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κέλλη, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς να εκφράσω την ε, συμπάθειά μου και αυτή της Ιρλανδικής κυβέρνησης για την καταστροφή της ε, συμβολικής Παναγίας των Παρισίων. Τώρα, για το Brexit τόσο τραβάει, τόσο περισσότερο υποφέρει ο κόσμος και δυστυχώς αυτό ισχύει για τις επιχειρήσεις που επηρεάζονται από το Brexit και για τους γεωργούς ε, που παίρνουν 100-200 ε, ευρώ ε, λιγότερα αναζώ από ό,τι πέρυσι, ακριβώς λόγω αυτής της αβεβαιότητας του Brexit. Ελπίζω λοιπόν ο Τερέζα Μέι και ο Τζέρμι Κόρμπιν να φτάσουν σε μια συμφωνία, αλλά πολύ αμφιβάλλουμε. Εάν όχι, θα πρέπει να ληφθεί μια απόφαση για να αναβληθεί το Brexit επάπειρον. Θα πρέπει να ε, υπάρξει βεβαιότητα. Επίσης επηρεάζεται η περιφέρειά μου γιατί πρέπει να εκλεγούν πέντε μέλη στην Ευρωκοινοβούλια, ενώ τώρα φαίνεται πως θα εκλέξουμε μόνο τέσσερις. Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε μόνο τους Βρετανούς γι' αυτό. Εγώ πριν από δύο χρόνια ζήτησα να μην δοθεί καμία έδρα μέχρι ότου να φύγουν οι Βρετανοί γιατί είχα πει ότι υπάρχει πιθανότητα να μην φύγουν μέχρι τις 29 Μαρτίου. Δυστυχώς βγήκα αληθινός. Ε, ε, εάν δεν ληφθεί απόφαση λοιπόν ε, για συμφωνία εξόδου θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Ευχαριστώ. Κάτσε διάει ο κύριος Ρανζέλ ένα λεπτό. Πρόεδρε, εγώ ήθελα να πω ότι με χαρά βλέπω πως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί έδειξαν ευελιξία με το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως είχαμε ζητήσει. Με χαρά βλέπω επίσης ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι διαθέσιμο για να οργανώσει ευρωεκλογέ και άρα ότι υπάρχει κάποια ε, πιθανότητα ο Βρετανικός λαός στο μέλλον να αποφασίσει να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως ε, θα ήθελα να είναι σαφές ε, ότι αυτή η απόφαση εξακολουθεί να δημιουργεί μεγάλη αστάθεια για τους ε, ανθρώπους, για τις εταιρείες και για τα κράτα ίδια. Γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τις εθνικές κυβερνήσεις να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους ώστε να ε, μπορέσουν να δώσουν ε, ε, βεβαιότητα στον κόσμο που υποφέρει λόγω αυτής της αναποφασιστικότητας του Βρετανικού Κοινοβουλίου και των αποφάσεών του. Κυρία Γκόμες, ένα λεπτό. Όλοι μας θρυνούμε για τη Γαλλία, για την ανθρωπότητα, γιατί η Παναγία των Παρισίων έχει χτιστεί από την ανθρωπότητα και η ανθρωπότητα θα την ξαναχτίσει. Θα ήθελα να πω πως λυπούμε πως το Συμβούλιο δεν έθεσε στην ημερήσια διατηξή για τη Βρετανία την υποχρέωση να ζητήσει ψήφο από τον λαό. Είναι ο δημοκρατικός τρόπος για να λυθεί αυτό το μπάχαλο, να αποφευθεί η Βρετανία να φύγει από την, Ευρωπαϊκή Ένωση και πιστεύω πως πλέον αυτό το μήνυμα θα πρέπει να σταλεί στο Βρετανικό λαό, στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, στα Βρετανικά κόμματα από τους ηθήνοντες στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι επίσης θα αντιμετωπίσουμε και τα αίτια της αποξένωσης των πολιτών που, οποίο οφείλεται το Brexit αλλά και ε, δείχνει ότι αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μεταρρυθμιστεί και να ξαναχτιστεί. Ευχαριστώ κυρία Μιράντα. Ένα λεπτό παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτή την Κυριακή πήγα στο Λονδίνο και μαζί με ένα σύλλογο Γαλλικιανών που είναι πολύ άριθμοι και ζουν στον Ηνωμένο Βασίλειο και υπάρχει αβεβαιότητα για την ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων, των υπηρεσιών και αβεβαιότητα επίσης για τα θέματα των ε, ε, ε, συνεπειών. Εργάζονται και ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι Ευρωπαίοι και Ευρωπαίες και δεν ξέρουν τι θα γίνει. Θέλω να πω επίσης, Πρόεδρε, και πρόεδρε Γιούνκερ για την πολιτική της αλληλείας των υπηρεσιών με βάση τα όσα γίνονται εδώ, με το τέλος αυτής της θητείας, είναι δικιά μας υποχρέωση να δείξουμε ευελιξία για να μπορέσει ο κόσμος που ζει στον Ηνωμένο Βασίλειο και που είναι Ευρωπαίοι να ε, ζήσει με μεγαλύτερη βεβαιότητα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Λόπες Αγγιγιά. Ευχαριστώ. Πρόεδρε η Ευρώπη πρέπει να περάσει σε άλλα θέματα. Πρέπει να συνεχίσει να βαδίζει προ τα μπρο και να επικεντρωθεί επιτέλου μετά από όλη αυτή την παγίδα του Brexit σε άλλα θέματα, για παράδειγμα, βλέπουμε πόσο θλιβόμεθα από την καταστροφή στο Νότρο Ντάμ. Στις 26 Μαΐου έχουμε μια υπαρξιακή σημασία εκλογική διαδικασία. Αλλά αντιμετωπίζουμε όλο και περισσότερες αβεβαιότητες για την σύνθεση και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γιατί έχει να κάνει με το αν θα συμμετάσχει όχι το Βασίλειο. Αναμένω λοιπόν να υπάρξει μία ε, απάντηση. Όχι μόνο δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία στη Βουλή των Κοινοτήτων, αλλά είναι πραγματικά απαράδεκτα ελαφρύ. Εδώ και 20 χρόνια καταδικάζουν ε, το ευρωπαϊκό εγχείρημα και επιτέλους περιμένω στις 26 Μαΐου οι φιλοευρωπαϊστές να συντρίψουν αποφασιστικά την δημαγωγία και την ευρωβαβία όχι μόνο στην, ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπρένον. Έχει περάσει η ώρα και μας μένει λίγος χρόνος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οικοδομήθηκε με βάση την εμπειρία από τον εφιάλτη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πόλεμου και ένας οραματισμός λόγω αυτού του πολέμου μας οδήγησε στην κατάσταση όπου είμαστε σήμερα. Και συμφωνώ λοιπόν με τα σχόλια του Πρόεδρου Τάσκ. Χρειαζόμαστε ακόμη ονειροπόλους. Όπως είπε και ο Τζι Λόρενς, όλοι ονειρεύονται, αλλά όχι με τον ίδιο τρόπο. Όσοι ονειρεύονται τη νύχτα στο υποσυνείδητό τους, ξυπνάνε τη μέρα για να βρουν ότι ήταν ματαιοδεξιό όλα αυτά. Αλλά όσοι ονειρεύονται μέσα στη μέρα είναι επικίνδυνοι, γιατί μπορεί να επιχειρήσουν ε, με ανοιχτά μάτια να καταστήσουν πραγματικότητα τα όνειρά τους, γιατί είναι αργά και μας μένει λίγος χρόνος. Πρόεδρε Τάσκ, σας καλώ να συνεχίσετε να ονειρεύεστε, να ονειρεύεστε κι εσείς που είστε κατά της παραμονής, αλλά να μην ονειρεύεστε απλώς, να κάνετε πραγματικότητα τα όνειρά σας. Μπορούμε να παραμείνουμε. Θα παραμείνουμε. Κύριος Χακμάρκ. Νομίζω ότι όλη η συζήτηση καταδεικνύει το εξής. Πόσο ισχυρή είναι η Ευρωπαϊκή Ενότητα. Τα προβλήματα στο Westminster δημιουργούνται από το ότι η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει πολλά για μια κοινωνία. Και είναι δύσκολο να ε, διαραγούν αυτοί οι δεσμοί. Και είμαι ευγνώμων που ο κύριος Φάραντζ είναι αστείος. Αλλά είναι απλώς αστείος. Ποτέ σοβαρά δεν έχετε συμβάλει στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, στην οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης, στο άνοιγμα των αγορών στην Ευρώπη. Απλώς ήσασταν αστείος. Γιατί να σας φοβόμαστε. Προσπαθείτε να μας φοβήσετε λέγοντας ότι θα ξαναγυρίσουμε εδώ. Μα κοιτάξτε, είστε απλώς ο γελοτοποιός ε, στην αυλή αλλά δεν χρειάζεται να σα ακούμε. Αυτά που λέτε δεν έχουν καμία έννοια για την ενότητα ή για του ε, λαού τη Ευρώπη. Είστε απλώ αστείο. Δεν σα φοβόμαστε. Και ελπίζω το Ηνωμένο Βασίλειο να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώνω τη διαδικασία Catch the Eye. Να δώσω το λόγο τώρα στον πρόεδρο Γιούνκερ. Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, Παίρνω τον λόγο. ώστε να ευχαριστήσω τους βουλευτές τώρα από αυτά τα χρόνια που ερχόμαστε στο Στρασβούργο όλοι. Θα είμαι παρόν και στην έναρξη των εργασιών του Προσεχούς Κοινοβουλίου, αλλά θα μου λείψει ο καλός φίλος Έλμαρ Μπροκ. Όλα αυτά τα χρόνια δουλέψαμε μαζί. Τσακωθήκαμε, συμφιλιωθήκαμε, γελάσαμε, πότε πότε κλάψαμε κιόλας. Ήταν τόσο ωραίο που συνεργαστήκαμε μαζί, Έλμαρ Μπρο, και σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε Γιούνκερ, ο Πρόεδρος Τούσκ. Μια παρατήρηση μόνο, Πρόεδρε. Πολλές εβδομάδες τώρα. έχει προξενήσει έντονες αντιδράσεις στο ενδεχόμενο συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στις ευρωεκλογέ. Θέλω να υπενθυμίσω προς άπασα κατεύθυνση πως το Ηνωμένο Βασίλειο έχει και δικαίωμα και υποχρέωση να λάβει μέρος στην εκλογική αυτή αναμέτρηση όσο είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό δεν είναι διαπραγματεύσιμο. Επίσης, δεν δέχομαι να ε, εγκαθιδρυθεί δεύτερη κατηγο... δεύτερης κατηγορίας συμμετοχή κράτους μέλους. Αντιλαμβάνομαι ότι ορισμένα ε, κομματικά συμφέροντα μπορεί να επισκιάζουν ή να επιχειρούν να επισκιάσουν την νομιμότητα. Ο κύριος Φερχόφστατ ε, επικροτήθηκε ενθουσιοδός από τον κύριο Φαράζ. Αυτό, κύριε Φερχόφστατ, θα έπρεπε για σας να αρκεί ως λόγος να αλλάξετε στάση και να διατυπώσετε με διαφορετικό τρόπο τα επιχειρήματά σας. Σας ευχαριστώ. Thank you. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ. Ολοκληρώνεται έτσι η συζήτηση.